τρίο και σε αυτήν συμμετέχει και η χώρα μου, η Κροατία και είμαι πεπισμένη ότι θα συνεργαστούμε επαρκώς. Είδα προσεκτικά το πρόγραμμα εργασίας σας και είμαι σίγουρη ότι τα ζητήματα συνοχής ε, θα σας απασχολήσουν πάρα πολύ. Επίσης για αυτό το οποίο είπατε για την σύνδεση και τη γεφύρωμα του καινού Βόρειας και Νότιας Ευρώπης ε, και επίσης η ασφαλής Ευρώπη την οποία αναφέρατε είναι κάτι το πολύ σημαντικό και πρέπει και η Ρουμανία και η Βουλγαρία και η Κροατία να μπουν στο χώρο Σέγγεν. Ελπίζω λοιπόν να μας βοηθήσετε για να μην έχουμε μια Ευρώπη δύο ταχυτήτων. Επιπλέον ε, στις προτεραιότητά σας ε, συμπεριλάβατε και την ισχυρή Ευρώπη που θα είναι ένας παγκόσμιος εταίρος. Βεβαίως αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Με ανησυχεί επίσης αυτό το οποίο είπατε ως τελευταίο σημείο την Ευρώπη των κοινών αξιών. Βεβαίω, υπάρχουν διάφορα ζητήματα εδώ πέρα, τα ακούσατε από τους συναδέλφους, υπάρχουν πολλές διαμαρτυρίες, πολλές διαδηλώσεις, ε, δυσαρέσκεια στους δρόμους και στη Ρουμανία σε εσά μάλιστα ίσως ε, αμφισβητείτε και το κράτος δικαίου. Και είπατε ότι πρόκειται βεβαίως για ένα ζήτημα επικουρικότητας. Έχετε ακούσει το τι φωνάζουν οι πολίτες στους δρόμους της ε, Ρουμανίας. Τους έχετε ακούσει όντως και θα τα εφαρμόσετε αυτά τα οποία ζητάνε. Και θέλετε να υπερασπίσετε το κράτος δικαίου στην χώρα σας. Αυτό έχει σημασία. Σας ευχαριστώ, Ροντρίκες. Welcome, ε, ήρθατε κυρία Πρωθυπουργέ. Η Προεδρία της Ρουμανίας θα είναι η πρώτη Προεδρία της χώρας σας. Και η τελευταία πρώτη της ευρωεκλογής. Και θα ήθελα τώρα να εστιάσω στην Σύνοδο Κορυφής του Σιμπίου που είναι η τελευταία μας ευκαιρία για να παρουσιάσουμε μια άλλη Ευρώπη για όλους τους πολίτες στην Ευρώπη πριν από τις ευρωεκλογέ. Να σας πω λοιπόν τι προσδοκούμε εμείς από εσάς για το τι είδους Ευρώπη θέλουμε εμείς μέσω της ε, Συνόδου Κορυφής του Συμπίου. Θεωρούμε ότι έχετε τις σωστές προτεραιότητες για να έχουμε ενότητα μεταξύ των Ευρωπαίων, συνοχή και οπωσδήποτε εδώ πέρα ε, η συνοχή είναι η λέξη κλειδί. Όπως είπατε, οικονομική, κοινωνική, πολιτική συνοχή. Είμαστε στο πλευρό σα. Και βεβαίω μπορεί να γίνει κάτι το πολύ συγκεκριμένο. Ο κοινωνικός πυλώνας να γίνει ευρωπαϊκό δίκαιο. Δεύτερον, μία πρώτη συμφωνία για τον πολιετή προϋπολογισμό όπου θα έχουμε ως κύρια ανησυχία την συνοχή θα περιλαμβάνει τα κρατη και την Ευρωζώνη. Και βεβαίως, ναι, να έχουμε μια Ευρώπη που θα βασίζεται στα ε, ευρωπαϊκά σύνορα και με την Ρουμανία. Το πρώτο είναι ακριβώς αυτή η συνεργασία με όλες τις σχετικές ε, χώρες. Το περιλαμβάνει και την ανατολική εταιρική σχέση που σας απασχολεί πάρα πολύ. Και βεβαίως αν τα καταφέρουμε σε αυτό θα μπορέσουμε να διαχειριστούμε και τη μετανάστευση. Και τέλος, ε, αν έχουμε αυτήν την Ευρώπη, θα έχουμε και ενότητα εότι και αν γίνει ιστορικό λοιπόν καθήκον, αλλά και μια ευκαιρία που έχετε. Ο κύριος Ντίβα, για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, η Ρουμανική Προεδρία είναι κάτι το οποίο μας καθησυχάζει, είμαστε σε καλά χέρια για το Brexit. Θέλω να μας βοηθήσετε σε αυτό. Πριν από δύο χρόνια θεωρούσαμε ότι θα είναι κάτι εύκολο το Brexit. Σήμερα είναι κάτι το οποίο όλοι θέλουν να ξεφορτωθούν. Και είναι δύσκολα τα πράγματα για την Πρωθυπουργό, την κυρία Μέη, η οποία πραγματικά έσφιξε τα δόντια και κάνει ό,τι μπορεί. Στη Βουλή των Κοινοτήτων απόψε θα γίνει χαμός. Αλλά βεβαίως η Πρωθυπουργό μας ε, δεν θα αλλάξει πορεία στη μέση του δρόμου. Ξέρει πως τα πράγματα είναι ζόρικα, αλλά θα κάνει ό,τι μπορεί για την Βρετανία. Ε, βρίσκεται βεβαίω μεταξύ σφύρας και άκμονος, αλλά αναμένουμε με κομμένη την ανάσα για κάποια επιτυχία. μινούτο. Ο κύριος Ζαντόφσκι για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να ευχηθώ ιδιαίτερα αποτελεσματική προεδρία στην Ρουμανία. Πολλά είναι αυτά που πρέπει να γίνουν, διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό, τους ε, νέους σχεδιασμούς της μεταναστευτικής πολιτικής, Υπάρχει μια σειρά δράσεων που προβλέπονται στο πρόγραμμα της Προεδρίας. Επίσης, η πολιτική συνοχή αποτελεί προτεραιότητα, πολύ σημαντική για μένα και είμαι σίγουρος ότι η Ρουμανία θα δώσει μια γεωπολιτική χρειά. Πρέπει να δούμε τι γίνεται και στα ανατολικά της Επίρου μας και σε σχέση με τη Ρωσία. Βέβαια, οι κύριες αξίες, ο σεβασμός του κράτους δικαίου είναι κάτι πολύ σημαντικό, αλλά νομίζω ότι πρέπει να ευχηθούμε στη Ρουμανία να μπορέσει να ξεπεράσει τα εμπόδια. Υπάρχει μια ερώτηση για σας, δέχεστε, παρακαλώ, κυρία Νικολάη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αναμφισβήτητα, η εκπεριτροπής Προεδρία θα είναι μια προκλητική Προεδρία. Δεν είναι εύκολο να μιλήσεις για το μέλος της Ευρώπης ε, όταν ε, παράλληλα τρέχει το Brexit. Όμως είναι πολύ εύκολο για κάποιους να μιλούν εκτός πραγματικότητας. Και αυτή η παραπληροφόρηση και η έλλειψη συνοχής ε, στο να κάνουν κάποιες δηλώσεις ε, είναι μία από τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναμφισβήτητα το κράτος δικαίου αποτελεί προτεραιότητα για τη Ρουμανία και αυτό το φαίνεται... Πρέπει να κάνετε μια ερώτηση, λέει ο Πρόεδρος. Μια ερώτηση πρέπει να θέσετε στον προηγούμενο μιλητή, στον κύριο Γιονταστόφσκι. Είμαστε δύο Νικολάη, κύριε Πρόεδρε. Ποιο μπορεί να μιλήσει. Ζητήσατε το λόγο. Για μπλε κάρτα. Θέλετε να θέσετε μια ερώτηση. Okay. Euh, Αν δεν έχετε ερώτηση, όχι, δεν έχω ερώτηση. Ε, μετά θα σας δώσουμε το λόγο τότε. Uh, Ο κύριος ε, Χόκμαρκ, παρακαλώ, για ένα μισή λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρωθυπουργέ, νομίζω ότι είναι φανταστικό το ότι η Ρουμανία αναλαμβάνει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, αυτό είναι ένα σημάδι για το πώς ε, έχει αναπτυχθεί η Ευρώπη. Όμως σίγουρα θα είναι φανταστική η εξέλιξη και θέλω να πω ότι εσείς και η δική σας κυβέρνηση πρέπει να καταπολεμήσετε τη διαφθορά όπως απαιτούμε και από οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση. Το να συγχωρείτε διεφθαρμένους πολιτικούς επειδή λέγεται ότι είναι, υπάρχει υπερπληθυσμός στις φυλακές δεν είναι αποδεκτό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το να καταπολεμάτε όσους καταπολεμούν τη διαφθορά είναι απαράδεκτο. Η αποποινικοποίηση της διαφθοράς, η, η αμνίστευση διαφθαρμένων για να προστατεύσετε τους δικούς σας δεν είναι αποδεκτό. Άκουσα ότι ο Ντο Μπούλμπαν σας υπεράσπισε, επικεφαλής σοσιαλιστικής ομάδας. Όμως αυτό είναι ντροπή για τη σοσιαλιστική ομάδα, πρέπει να πω. Υποτίμησε τον εαυτό του και εσείς θα πρέπει να αναλάβετε την ευθύνη να προστατεύσετε τη Ρουμανία γιατί πιστεύουμε ότι είναι φανταστικό το ότι έχετε αναλάβει την Προεδρία αλλά μην τα θαλασσώσετε. Έχετε μια ευθύνη και πρέπει να την αναλάβετε. Κύριε Χόκμαρκ, υπάρχει μπλε κάρτα για σας, δέχεστε, από τον κύριο Φρουντσουλίκα. Παρακαλώ, η ερώτησή σας. αγαπητέ συνάδελφοι. Δεν πιστεύετε ότι είναι ντροπή σήμερα ο πρόεδρος ε, του ΕΛΚ, ο κύριος Σοζουφτόλ, συνεχάρει τον κύριο Γιωχάνης και του είπε ότι θα ε, υλοποιήσει μια εξαιρετική προεδρία όταν ξέρουμε όλοι ότι την εκπεριτροπής προεδρία του Συμβουλίου την αναλαμβάνει η κυβέρνηση της Ρουμανίας και επικεφαλής είναι η Ρουμάνα Πρωθυπουργός. Δεν είναι λοιπόν ντροπή ο κύριος Κούρς στις 21 Δεκεμβρίου του Βουκουρέστη, στο Βουκουρέστι παρέδωσε συμβολικά την Προεδρία του Συμβουλίου στον πρόεδρο Γιωχάνης, κάνοντας εκ νέου ένα μεγάλο πολιτικό λάθος. Και ταυτόχρονα ε, ουσιαστικά παραπλάνησε τους πολίτες που πρέπει να ξέρουν την αλήθεια. Παρακαλώ να απαντήσετε. Κύριε Πρόεδρε. Πιστεύω ότι κάπου έφυγε εκτός θέματος ο συνάδελφος, γιατί εγώ μιλούσα για τα προβλήματα της διαφθοράς στη Ρουμανία. Όπως ε, μας έχει καταδείξει η Transparency International, η Επιτροπή της Βενετίας και πολλοί άλλοι. Και το γεγονός της αμνίστευσης ε, διεφθαρμένων πολιτικών και μόλι μίλησε ο υπουργό ε, στο BBC. Είπατε ότι κάποιοι δίνουν τα συγχαρητήρια στον πρόεδρο της χώρας σας. Ε, τι να σας πω, εμένα δεν με ανησυχεί και πολύ αυτό. Νομίζω ότι εσείς και οι σοσιαλιστές εδώ θα πρέπει να, είναι, να είστε τόσο αυστηροί με τη Ρουμανία όπω είμαστε και με την Ουγγαρία ή την Πολωνία. Γιατί η κατάχρηση εξουσίας πάντοτε είναι κατάχρηση εξουσίας. Θα πρέπει και εσείς και εμείς να την καταπολεμήσουμε. Κυρία Φαγιόν, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρία Πρωθυπουργέ, στην αρχή της Προεδρίας σας έχετε προσελκύσει ήδη μεγάλη προσοχή. Πιστεύω, ωστόσο, ότι θα πετύχετε τους στόχους σας στη διάρκεια της Προεδρίας σας. Εγώ σας υποστηρίζω, ιδίως ό,τι αφορά τα Δυτικά Βαλκάνια. Θα πρέπει να δείξουμε θετική κά παραδείγματα ε, σε αυτήν την περιοχή της Ευρώπης και γι' αυτό ε, συγχαίρω τους φίλους μας ε, στην Μακεδονία που ψήφισαν υπέρ των συνταγματικών αλλαγών. Και η Ελλάδα πιστεύω ότι θα ψηφίσει θετικά. Ήταν πραγματικά τολμηρό και σοφό εκ μέρους των ηγετών να επιδιώξουν την επίλυση αυτής της διαφιλονικίας. Καλό λοιπόν τους ηγέτες της περιοχής και την Προεδρία να εξομαλύνουν με μεγάλη αυστηρότητα ε, την κατάσταση. Να μην υπάρχει μίσο και καχυποψία κατά των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Χρειαζόμαστε ενωμένη Ευρώπη, η οποία θα έχει και κοινωνική διάσταση. Θέλουμε να είναι σταθερή και ειρηνική. Εύχομαι να οδηγήσετε εσεί την Ευρώπη σε αυτή την πορεία. Ευχαριστούμε. Τόμας, έτσι για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η Ρουμανία αναλαμβάνει για πρώτη φορά την Προεδρία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε ένα διάστημα χρονικό ιδιαίτερα δύσκολο. Θα πρέπει να επικεντρωθείτε στο πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο και να λάβετε υπόψη και την απώλεια ενό του κράτου μέλου, μαζί με τι ευρωεκλογέ που θα καθορίσουν το μέλλον τη Ένωσή μα. Ελπίζω λοιπόν ότι τα εσωτερικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ρουμανία δεν θα πλήξουν και τι φιλοδοξίε τη, όπω τι έχει εκφράσει στο πρόγραμμα προτεραιοτήτων τη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να χάσει χρόνο, διότι για να επικεντρωθούμε στι οικονομικέ μα προτεραιότητε θα πρέπει να βιαστούμε. Ούτε τι μεταναστευτικέ προκλήσει μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αργότερα, γιατί από εμά περιμένει μια ε, θαραλέα κίνηση ο υπόλοιπο κόσμο. Ελπίζω λοιπόν η Ρουμανική Προεδρία να ε, ασχοληθεί με την επίλυση αυτών των προβλημάτων όπω έχει ανακοινώσει. Και η ασφάλεια δεν θα πρέπει να ε, γίνει μια ε, πουσιώδη προτεραιότητα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι τόσο ασφαλή όσο ήταν στο παρελθόν. Αυτό το αποδεικνύουν οι πολλαπλέ απόπειρε. Θα πρέπει να δώσουμε μεγάλη έμφαση στην ασφάλεια των προτεραιοτήτων μα. Ο κ. Μαρινέσκου. Ευχαριστώ. Είναι πολύ μεγάλη ικανοποίηση για μένα να μπορώ να διαπραγματεύομαι τα νομοθετήματα με την Ρουμανική Προεδρία. Εγώ έχω την εξή θέση ως μέλος του ΕΛΚ. Εργάζομαι ήδη και θα εργαστώ με τη μόνιμη προσωπία της Ρουμανίας και θα συνεισφέρω στο να κλείσουν νομοθετικοί φάκελοι. Θα συνεχίσω να υπερασπίζω τα συμφέροντα των Ρουμάνων σε όλους ε, τους φακέλους ε, που είναι σε εξέλιξη. Δεν δέχομαι θέσεις ε, κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εγώ θα θα καταφερθώ κατά θέσεων που αφορούν τον περιορισμό της κυκλοφορίας των εργατών. Κυρία Ντανσίλα, Μιλήσατε πολύ για την πολιτική συνένεση σε εσωτερικό επίπεδο. Εγώ δεν ε, συμφωνώ με τέτοια συνένεση κατά των ευρωπαϊκών αξιών του κρατού δικαίου και τη δικαιοσύνη. Ε, ζητήσατε ένταξη στο χώρο Σενγκεν. Δεν είναι πολύπλοκο. Διορθώστε του νόμου περί δικαιοσύνη. Ε, στείλετε του υπουργού να συζητήσουν στι ευρωπαϊκέ πρωτεύουσε και να πείσουν τι κυβερνήσει να ψηφίσουν υπέρ τη Ρουμανία. Και ε, όποιον στείλετε θα προεδρεύσει και του Συμβουλίου Δικαιοσύνης. Χρησιμοποιήστε τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Η Ρουμανία χρειάζεται νοσοκομεία, δρόμους, σιδηροδρομικές γραμμές. Αν κάνετε όλα αυτά θα δείξετε ότι είστε στην πλευρά των Ρουμάνων και θα κερδίσετε το σεβασμό των Ευρωπαίων εταίρων. Η υποχρέωσή σας είναι να εκπροσωπήσετε τη Ρουμανία σύμφωνα με την επιθυμία της ε, πλειοψηφίας ε, των πολιτών και όχι σύμφωνα με την πλειοψηφία των βουλευτών ε, του. Έχετε μία μπλε κάρτα, τη δέχεστε. Ο κύριος Γιακονσάρη, παρακαλώ, κάντε την ερώτηση. Η κυρία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αναρωτιόμουν για το ότι κανείς δεν μίλησε για μία από τις ε, μεγαλύτερες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρώπη που λαμβάνει η χώρα στη Ρωμανία, δηλαδή τους Ρωμά και τη μεταχείρισή τους. Και εσείς ε, είστε Πρωθυπουργό, Θα ήθελα λοιπόν να σα ρωτήσω μήπως αυτό οφείλεται ότι τα πράγματα έχουν βελτιωθεί ή συχνά σε τέτοιες συζητήσεις είμαστε τόσο ευγενικοί και δεν θίγουμε τα δύσκολα. Σας ευχαριστώ ο κύριος Μαρνέσκου για να απαντήσει. Είναι μία ερώτηση που προέρχεται από έλλειψη σωστής ε, ενημέρωσης. Ε, σας καλώ να έρθετε στη Ρουμανία και στη δική μου περιφέρεια, όπου ήρθαν ε, και άλλοι συνάδελφοι, να επισκεφτείτε την πόλη και την περιοχή σας. Καλό να αλθείτε και να δείτε τι συμβαίνει σε σχέση με το θέμα που θίξατε εδώ στη Ρουμανία. Ευχαριστούμε ο κύριος Βάιντεν Χόλτσερ. Γιώζεφ, ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Κυρία Πρωθυπουργέ, κάθε χρόνο αλλάζει η Προεδρία του Συμβουλίου. Είναι δηλαδή κάτι το σύνηθες σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η ανάληψη της ε, Προεδρίας από τη Ρουμανία αποκλίνει αυτό το, από αυτό το σχήμα γιατί αφενός ε, υπάρχει ιδιαίτερη χρονική πίεση και από την άλλη ε, όλη η χώρα πλέον ε, είναι υπό το μικροσκόπιο ολόκληρη της Ευρώπης. Ε, η Κομισιόν πριν από λίγες εβδομάδες διαπίστωσε μια στασιμότητα όσον αφορά την κατάσταση του κράτους ε, δικαίου στην χώρα. Η Ρουμανία λοιπόν θα βρεθεί υπό το μικροσκόπιο του επόμενου μήνε. Και εδώ πέρα υπάρχει μια ευκαιρία. Η χώρα μπορεί να δείξει ότι είναι ικανή να επιλύσει τα εσωτερικά τη προβλήματα και τι υποχρεώσει ε, που έχει. Είμαστε πεπισμένοι ότι μπορεί να επιτύχει πολλά η Ρουμανία σε ευρωπαϊκό επίπεδο και θα σα στηρίξουμε σε αυτό. Σα ευχαριστώ, Γιώζεφ. Κύριο Γιούρεκ, για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πριν να χρησιμοποιήσω το λεπτό μου θα ήθελα να πω ότι ο κύριος Μπούλμαν πριν 20 λεπτά παρενέβη. Εγώ τότε είχα ζητήσει να πάρω το λόγο γιατί ήθελα να αφιστήσω την προσοχή του Προέδρου Ταγιάννη. Το άρθρο 11 του κανονισμού μας υποχρεώνει στο να σεβόμαστε ο ένας τον άλλο και να μην προβαίνουμε σε δηλώσεις δυσφημιστικές. Τώρα, πρόκειται για μια κυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναφέρθηκε ως φασιστική. Ε, εδώ μιλάμε για ε, μία από τις μεγαλύτερες ομάδες αυτού του κοινοβουλίου να επιτίθεται σε αυτή την κυβέρνηση. Δεν είναι παραδεκτό αυτό. Ο πρόεδρο έπρεπε να έχει αντιδράσει αμέσω. Και όταν ένας βουλευτής ζητά το λόγο, δεν ε, είναι δυνατό να μην δίνεται το λόγο για ένα διαδικαστικό ζήτημα. Ο κύριος Μπούλμαν δεν είναι ο μόνος που έχει δικαίωμα να αντιδρά στις παρεμβάσεις άλλων συναδέλφων. Γι' αυτό εγώ θέλω να εφιστήσω την προσοχή, εφιστήσω την προσοχή του Πρόεδρου Ταγιάννη στο γεγονός αυτό. Τώρα, σε σχέση με την απάντηση του κυρίου Μπούλμαν, δεν υπήρξε αντίδραση από την πλευρά του Προέδρου και Τώρα να περάσω και στη δική μου παρέμβαση. Τώρα αρχίζει να μετράει το δικό μου λεπτό. Συγγνώμη. Εσείς πήρατε το λόγο για ένα θέμα που έχει να κάνει με τον πρόεδρο Ταγιάννη που ήταν εδώ στην αίθουσα και ξέρει πάρα πολύ καλά το ζήτημα. Εγώ θα του το παραπέμψω. Όμως αυτό έχει να κάνει με τη δική του παρέμβαση. Παρακαλώ. Κύριος Ανδρία, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, κυρία Πρωθυπουργέ. Ευχαριστούμε που ήρθατε σήμερα το απόγευμα. Ήθελα να μιλήσω σήμερα για το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο με την ευκαιρία τη επισκεψή σα. Όπω ξέρετε, η θέση του Κοινοβουλίου εδώ είναι ξεκάθαρη. Χρειάζεται ένα επίπεδο δαπανών φιλόδοξο, το οποίο να ασχολείται με την υλοποίηση των στόχων τη βιώσιμη ανάπτυξη, ξεκινώντα από την καταπολέμηση τη υπερθέρμανση του πλανήτη και των κοινωνικών ανισοτήτων καθώ και των εδαφικών. Ε, εδώ βλέπουμε να αναδαβλίζονται οι, μάλλον οι εξτρεμισμοί, να κινδυνεύει το ευρωπαϊκό εγχείρημα και η οικονομική μα σταθερότητα. Πρέπει το Συμβουλίο να καταλάβει ότι χωρί αυξήσει στου ίδιου πόρου, το Κοινοβούλιο δεν θα μπορέσει να δώσει τη συνένεσή του για την διάσταση των δαπανών. Θα πρέπει λοιπόν και για του πόρου να δείτε ότι είναι μηδενική η πρόοδό μα. Θα πρέπει να δούμε τι αδρέ γραμμέ ε, πιθανή συνεννόησή μα για τι ε, δημοσιονομικέ γραμμέ. Τι εννοείται από τη μια μεγάλε γραμμέ και από την άλλη πώ θα λάβετε υπόψη τι διαφορετικέ θέσει του Κοινοβουλίου στα διάφορα αυτά θέματα. Ευχαριστούμε, κυρία Μπρέσο. Παρακαλώ, Μερτσέντε, για ένα λεπτό. Πρόεδρε, κυρία Πρωθυπουργέ, και από μένα πολλέ ευχέ για καλή έκβαση στην Προεδρία σα. Ευχαριστούμε για τις τέσσερις θεματικές προτεραιότητες που μας ε, αναφέρατε. Θέλω να σχολιάσω το θέμα της εδαφικής σύγκλησης. Πιστεύω ότι καμία περιοχή της Ευρώπης, όπως θυμήσατε και εσείς, δεν πρέπει να μείνει ε, καθυστερημένο στην ε, πρόοδο που θα κάνουν οι υπόλοιποι. Γιατί, ε, όπως είπαμε εδώ στο Κοινοβούλιο πριν από κάποιο καιρό, Χρειάζεται ένα κατάλογο προτεραιοτήτων και για τι περιοχέ που έχουν καθυστερήσει αυτέ τι υπαίθρου, τι ορεινέ και τι εξόχω απόκεντρε περιοχέ. Όχι μόνο λοιπόν για τι αστικέ περιοχέ, αλλά και για αυτέ τι ε, απομακρυσμένε περιοχέ, τι μειονεκτούσε περιοχέ. Κατάλογο προτεραιοτήτων. Το έχει ζητήσει και το Κοινοβούλιο με μια πρωτοβουλία του. Πρωτοβουλία που ξεκίνησε μια πρώτη μελέτη του θέματο και θα μπορούσε μετά να οδηγήσει και σε εκπόνηση μια ε, τέτοια ε, ιεραράχηση των στόχων. Είναι σημαντικό λοιπόν η Προεδρία, γιατί η Ρουμανία είναι μια χώρα με πολλέ ε, περιοχέ υπαίθρου, αγροτικέ περιοχέ, ορεινέ περιοχέ στην Ευρώπη. Τα γνωρίζετε καλά. Ε, ένα δευτερόλεπτο ακόμα. Πάνω από ένα εκατομμύριο νέοι θα ψηφίσουν για πρώτη φορά στι ευρωεκλογέ φέτο. Τι σκέφτεστε να κάνετε για να συμμετάσχουν ενεργότερα και για να του εξυπηρετήσετε και να του βοηθήσετε μάλλον και να διευκολύνετε την έλευσή του στι κάλπε. Ευχαριστούμε κύριε Μπρέσο. Ε, κυρία Μπρέσο, κύριο Νίτσα. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρωθυπουργέ, αγαπητά μέλη της κυβέρνησης, καταρχήν θα ήθελα να σας ε, συγχαρώ που παρουσιάσατε τις προτεραιότητες και το πρόγραμμα δραστηριοτήτων της Ρουμανικής Προεδρίας. Και επίσης ε, θα ήθελα να σας ε, παρακαλέσω να μην μπερδευτείτε εδώ, επειδή το τι είπε κάποιος συνάδελφος εδώ δεν είχε καμία σχέση με την Προεδρία της Ρουμανίας, ούτε με το πρόγραμμα τα δραστηριοτήτων απλώ εντάσσεται στην προεκλογική εκστρατεία. Θα πρέπει να κατανοήσετε τον κύριο Βερχόφστατ. Ε, ε, δεν ε, φτάνει το αντίστοιχο κόμμα στην Ρουμανία στο εκλογικό κατόφλι και γι' αυτό γίνονται όλα αυτά. Ταυτόχρονα θέλω να σα ενθαρρύνω μαζί με του 200 υπαλλήλου τη μόνιμη αντιπροσωπεία τη Ρουμανία μαζί και με άλλου εκατοντάδε υπαλλήλου που στη Ρουμανία προετοιμάζουν την Προεδρία. Να ακολουθήσετε το χρονοδιάγραμμα παρουσίαση σε κυρία Πρωθυπουργό, γιατί οι τέσσερις πυλώνες, η σύγκληση, η ασφάλεια, η παγκόσμια Ευρώπη και η Ευρώπη των αξιών είναι ένα θέμα που θα μείνει στη Ρουμανία, στην ιστορία για τη Ρουμανία και θα θεωρηθεί ότι είναι το πιο πολιτικό σημαντικό βήμα που έκανε η Ρουμανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε και καλή επιτυχία κυρία Πρωθυπουργέ. Ευχαριστώ κυρία Νίκα. Η κυρία Τόια, παρακαλώ, έχει το λόγο για ένα λεπτό. Πρόεδρε, θέλω να χαιρετήσω την Πρόεδρο του Συμβουλίου σε αυτό το στάδιο. Είναι μια συνάδελφος που την εκτιμούσαμε στην ομάδα μας και στο Κοινοβούλιο. Θέλω να υπογραμμίσω κάποιες πτυχές γιατί αναφέρθηκαν πολλά από τους συναδέλφους της ομάδας μου και θέλω να αναφερθώ σε δύο σημαντικές στο, θέμα του κοινωνικού πυλώνα. Είναι ένας από τους τέσσερις πυλώνες ε, που παρουσίασε στο πρόγραμμά της η Ρουμανική Προεδρία και νομίζω ότι μπορεί να είναι ένα θέμα αξιολόγηση της δράσης και της ικανότητας της Ευρώπης σε αυτή την κρίσιμη εποχή για τους Ευρωπαίους πολίτες σε κάποιες ε, χώρες είναι πιο προφανής η κοινωνική προσοχή ε, που, της οποίας χρήζουν οι πολίτες μας, άλλες δεν είναι τόσο προφανής, όμως χρειαζόμαστε μια Ευρώπη που να ε, φροντίζει τα παιδιά και να προωθεί την ευημερία. Μία άλλη πτυχή είναι αυτή τη βιομηχανία. Εγώ τα βλέπω μαζί, γιατί μια αλλη πτυχη ειναι αυτη της βιομηχανιας εγω τα βλεπω μαζι γιατι μια ευρωπη που μεγενθύνεται είναι και μια Ευρώπη που μπορεί να είναι πιο κοντά στις ε, ανάγκες και σκέφτομαι και το πρόγραμμα Ορίζοντα, Horizon και εγώ νομίζω ότι η Προεδρία θα πρέπει να ολοκληρώσει με τη συνεισφορά όλων. Σας ευχαριστώ και καλή δουλειά. Ο κύριος Ντάντη για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κυρία Πρωθυπουργέ, Καλώς επιστρέψατε στην αίθουσα του Κοινοβουλίου, την αίθουσα της Ολομέλειας. Δεν έχετε πολύ χρόνο λόγω των ευρωεκλογών. Θα πρέπει να ασχοληθείτε με σημαντικά θέματα. Νομοθετική δουλειά σημαντική μαζί με το Ευρωκοινοβούλιο. Επειδή δεν υπάρχει πολύ χρόνο, θα σταθώ σε ένα σημείο που μου είναι ιδιαίτερα προσφυλέ. Το θέμα τη ενιαία αγορά. Όπω όλοι ξέρουμε, είναι μια μεγάλη, από τι μεγάλε επιτυχίε τη ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Δυστυχώ όμω έχει ακόμα πολλέ αδυναμίε. Και τα τελευταία χρόνια έχουν ε, υπάρξει φόβοι λόγω της ενίας αγοράς και αντιευρωπαϊκές τάσεις. Θα πρέπει λοιπόν να ορίσετε μια συγκεκριμένη οδό δράση, πορεία δράση μάλλον, με κανόνε αυστηρού για την ψηφιακή μετάβαση τη ε, κοινωνία και τη οικονομία μα. Και επ' αυτού να υπογραμμίσω το εξή. Ένα ακόμη θέμα τον κανονισμό για την εποπτεία της αγοράς. Ελπίζω μαζί με την Ρωμανική Προεδρία να μπορέσετε να ολοκληρώσετε τις διαγματεύσεις της προσεχής εβδομάδες. Πιστεύω ότι πρέπει να διασφαλίσουμε στους Ευρωπαίους πολίτες προϊόντα ασφαλή ιδίω αυτά που πολλούνται στο διαδίκτυο και σύμφωνα όλα με τα πρότυπα και του κανόνε μα. Είναι ε, σημαντικό για την εσωτερική αγορά και για να υπάρχει θεμητό ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων τη Επίρου μα. Ευχαριστούμε κυρία Ντάντη. Και τώρα για την διαδικασία Catch έχουμε 25 εγγεγραμμένου. Είναι αδύνατο. Δεν μπορώ να δώσω το λόγο σε όλου. Θα δώσω το λόγο σε 10 ομιλητέ. Ανά ομάδα για να μπορέσουν όλοι να λάβουν το λόγο. Κύριος Πασκού. Ένα λεπτό. Κυρία Πρωθυπουργέ, κύριε Πρόεδρε, κάθε Προεδρία θα πρέπει να δράσει πάνω σε τρεις γραμμές. Καταρχήν να συνεχίσει τις εργασίες της προηγούμενης Προεδρίας, δεύτερον να πετύχει τους δικούς της στόχους και τρίτον να ενταχθεί στο συγκεκριμένο πλαίσιο που βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Ένωση την αντίστοιχη στιγμή. Μα παρουσίασε το πρόγραμμα Ρουμανία, σεβόμενη αυτά τα αιτήματα. Σήμερα, όταν ε, η φιλελεύθερη τάξη ε, βρίσκεται σε κρίσιμη στιγμή, η Ρουμανία προτείνει μέσω τη Προεδρία τη να ενδυναμώνει την Ευρωπαϊκή Ένωση ω κύριο πυλώνα του συστήματο αυτού. Ταυτόχρονα, να μην ξεχνάμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει ισχυρή όχι μόνο ως ε, θεσμός αυτός καθ' αυτός, αλλά και χάρη στις προσπάθειες του κάθε κράτους μέλους. Στο σημερινό κόσμο και στον ευριανό κόσμο η προστασία που προβλέπεται από τα θεσμικά όργανα θα πρέπει να διπλασιαστεί και να υπάρχουν και οικονομικές και στρατιωτικές προσπάθειες από τα κράτη-μέλη παράλληλα με τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτούς ε, ε, ε, δεν μπορούμε να τους πετύχουμε μέσω της διάκρισης και την απομόνωση παρά μόνο αν υπάρχει ειλικρινή συνεργασία μεταξύ όλων των κρατών μελών. Ευχαριστώ κύριος Μουρεσάν για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Κυρία Πρωθυπουργέ, αγαπητοί συνάδελφοι, η ανάληψη τη Προεδρία του Συμβουλίου τη Ευρωπαϊκή Ένωση για πρώτη φορά είναι ιστορική στιγμή για τη χώρα μα και θέλω να πω ξεκάθαρα ότι η Προεδρία αυτή ανήκει καταρχήν στο ρουμανικό λαό. Και θέλω να πω επίση ξεκάθαρα, ο ρουμανικό λαό είναι έτοιμο για αυτή την πρώτη Προεδρία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Βλέπουμε ότι εδώ και δύο χρόνια διαδηλώνουν οι Ρουμάνοι είτε στο δρόμο για να υπερασπίσουν το κράτο δικαίου και μια ανεξάρτητη τη δικαιοσύνη και τις ευρωπαϊκές αξίες και το κάνουν κρατώντας ε, την σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όμως ε, ε, πέρα από το ότι αποτελεί τιμή αποτελεί και ευθύνη η Προεδρία και εσείς κυρία Πρωθυπουργή θα έχετε την δυνατότητα να διαχειριστείτε κάποια σημαντικά θέματα. Καταρχήν, τον προπολογισμό για τα επόμενα 7 χρόνια. Στου ε, δικαιούχου ε, θα πρέπει να δώσουμε βεβαιότητα ω προ τα ποσά ε, και ω προ τι προποθέσει βάσει των οποίων θα λάβουν χρήματα. Για τον Brexit θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει απόψε και θα πρέπει να προσφέρουμε στα εκατομμύρια Ευρωπαίου πολίτε που βρίσκονται στη Βρετανία βεβαιότητα για το μέλλον του. Τρίτον, η Ρουμανία έχει την ε, δυνατότητα ε, να θέσει την ανατολική Γετνία τη Ευρωπαϊκή Ένωση στο θεματολόγιο της Ευρωπαϊκής Ένωση. Όμως πρέπει να σέβεστε τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωση. Αυτό περιμένει η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ίδιο περιμένει και ο ρουμανικός λαός. σα. ευχαριστώ. Προσπαθήστε να σεβέστε το χρόνο, συνάδελφοι. Ο κύριος Μαριάς, για ένα λεπτό. Κυρία Πρωθυπουργέ της Ρουμανίας, εγώ θα αναφερθώ στο μεταναστευτικό γιατί είμαστε ξανά στο ίδιο έργο θεατές με το συμβούλιο να είναι ανίκανο να αναλάβει τις ευθύνες του καθώς συγκεκριμένα κράτη μέλη συνεχίζουν το business as usual και αρνούνται να αλλάξουν το δουβλίνο τρία που έχει μετατρέψει την ελλάδα και την ιταλία σε αποθήκες ψυχών. η ελλάδα δεν αντέχει πλέον άλλους πρόσφυγες και παράνομους μετανάστες. τα νησιά του αιγαίου έχουν βουλιάξει από τους μετανάστες και από τις αυξημένες ροές οι οποίες πλέον υπάρχουν και χερσαία στον εύρο. η περίφημη αλληλεγγύη της ευρωπαϊκής ένωσης παραμένει γράμμα κενό. πρέπει λοιπόν να εκτελεστεί η μετεγκατάσταση. έχει εκτελεστεί μόνο κατά το. 30%. προτείνω να αλλάξει το σύστημα χορήγησης ασύλου να καταργηθεί το δουβλίνο iii και η ρύθμιση του κράτους πρώτης εισόδου να γίνει κατανομή των αιτήσεων ασύλου καθώς και των προσφύγων και μεταναστών μεταξύ των κρατών μελών με βάση την έκταση τον πληθυσμό και το αεπ. έτσι θα εκφραστεί η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. περιμένουμε μέτρα από την προεδρία σας. ευχαριστώ όσους εκφράσατε την εμπιστοσύνη σας στην Ρουμανική Προεδρία και εγώ ήμουν μέρος της κυβέρνησης. Ξέρω πολύ καλά τα μέλη της κυβέρνησης και είμαι σίγουρη γιατί θα ασκήσουν μια καλή Προεδρία. Για πρώτη φορά είχαμε ένα διευρυμένο συμβούλιο και εμείς εργαστήκαμε ως ευρωβουλευτές για το πρόγραμμα. Έχουμε πολύ Έχουμε προετοιμαστεί πολύ καλά, όμως είναι λυπηρό που οι συνάδελφοί μας ε, που ήρθαν στο Κοινοβούλιο με ψευδείς πληροφορίες ε, όταν εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προσπαθούμε να εξελίψουμε τις ψευδείς ειδήσει. Ε, εντάξει, είμαστε τη προεκλογικής εκστρατεία, αλλά δεν πρέπει να επιτεθόμαστε σε ένα κρατός μέλο που αναλαμβάνει την Προεδρία. Πρέπει να μιλήσουμε για την προτεραιότητα, για το πρόγραμμα. Θα ήθελα να ρωτήσετε περισσότερο τι μπορούμε να κάνουμε κάνουμε, πώς, να προτείνετε προτεραιότητες, όχι να αρχίσουμε να μιλάμε για πράγματα που δεν ξέρουμε και σας διαβεβαιώ ότι δεν τα ξέρετε. Εγώ εύχομαι κάθε επιτυχία στην Προεδρία και μάλιστα σήμερα ψηφίστηκε στην Ολομέλεια ένα θέμα για το οποίο είμαι η συγγήτρια και θα ξεκινήσουμε τις οργανικέ διαπραγματεύσεις. Θα δείτε τι καλή Προεδρία λοιπόν θα ασκήσει η Ρουμανία. Συγχαρητήρια και καλή επιτυχία. Κυρία Κούνεβα, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητή κυρία Πρωθυπουργέ, χαίρομαι που σας ξαναβλέπω εδώ. Το 2018 συμμετείχατε ως ευρωβουλευτή, στην εκδήλωση που διοργανώσα με δύο συνάδελφους από την πολιτική σας ομάδα, τον κύριο Πυρίνσκι από τη Βουλγαρία και την κυρία Γκραπίνη από τη Ρουμανία, για να αναζητήσουμε νέους δρόμους συνεργασίας στα Βαλκάνια. Ελπίζω ότι τώρα θα πράξετε τα μέγιστα για να προχωρήσει η βαλκανική συνεργασία. ανησυχούμε όμως όταν ακούμε ότι η ρωμανία είναι ένα πολύ κακό παράδειγμα για τις εργασιακές σχέσεις τους μισθούς την κοινωνική ασφάλιση και τα δικαιώματα. είναι έτσι; τέσσερα χρόνια δουλέψατε μαζί μας και ξέρετε τις προτεραιότητες που έχει το ευρωκοινοβούλιο κοινωνικός πυλώνας ανθρώπινα δικαιώματα αναθεώρηση του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου. Αυτές πρέπει να είναι και οι δικές σας προτεραιότητες. Σας εύχομαι καλή προεδρία και να πάνε όλα με τον καλύτερο τρόπο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριος Γιάροκ για ένα λεπτό. Ή κυρία Γιάροκ. Κυρία ε, Πρωθυπουργέ, ευχόμαστε κάθε επιτυχία στην Προεδρία σας και σας ευχαριστούμε που τονίσατε τα κυριότερα σημεία. Ένα από τα σημαντικότερα για εμάς είναι η συνοχή την οποία αναφέρατε και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όχι μόνο όταν μιλάμε για τις οικονομικές διαφορές όπως είπατε α, μεταξύ των ανθρώπων αλλά και την πρόσβασή τους στα δικαιώματα ως Ευρωπαίοι πολίτες. Η κοινωνική και περιφερειακή συνοχή λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντική και αναμένουμε από εσάς να κάνετε κάτι τους επόμενους έξι μήνες γιατί θεωρούμε ότι έχετε μεγάλη πείρα σε αυτά τα θέματα. Ε, ε, έχετε, είστε σε ένα από τα πιο φτωχά κράτη-μέλη. Προσπαθείτε να αλλάξετε την κατάσταση. Σας ευχαριστώ για την ερώτηση για τους Ρωμά και την απάντηση κύριε Μαρινέσκου γιατί ξέρω γιατί υπόθηκε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξαναδούμε το θέμα των φτωχών. Νομίζω πως η Προεδρία σας πραγματικά πρέπει να στείλει ένα μήνυμα στην Ευρώπη πως ε, υπάρχουν 220 εκατομμύρια φτωχοί στην Ευρώπη που πρέπει να βοηθηθούν. Ελπίζω λοιπόν η Προεδρία σας να προωθήσει το θέμα αυτό. Σας ευχαριστώ λοιπόν. Σας ευχαριστώ. Ζωάννα παρακαλώ για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρο, κύριε Πρωθυπουργέ, αγαπητά μέλη, της κυβέρνησης Ρουμανία, Ρουμανίας, αγαπητοί συνάδελφοι, ίσως να μην είναι τυχαίο σήμερα ότι 12 χρόνια μετά την προσχώρηση της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση με την ευκαιρία της παρουσίασης των προτεραιοτήτων ε, της ε, Προεδρίας γιορτάζει δύο σημαντικέ επαιτίου στη Ρουμανία. 116 χρόνια από τη γέννηση του Μιχαέ Μινέσκου, του εθνικού μας σπίτι που έχει μεταφραστεί σε πάνω από 60 γλώσσες και την ημέρα ε, του εθνικού μας πολιτισμού. Για μας αυτό που συμβαίνει εδώ σήμερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όταν ε, η Ρουμανία μέσω της φωνής της κυρίας Δεντσίλα της Πρωθυπουργού, της Πρωθυπουργού παρουσιάζει το όραμά της ε, για την εντολή της Προεδρίας ε, αποτελεί μια τρίτη αιτία γιορτής. Μας κάνει να αισθανόμαστε περήφανοι γη και κόρες αυτής της μεγάλης οικογένειας. Και θέλω να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία για να ευχηθώ κάθε επιτυχία στην κυρία Νταντσίλα και στα μέλη της ρουμανικής κυβέρνησης και να παρακαλέσω τους συναδέλφους να έχετε εμπιστοσύνη στις ικανότητες και στο όραμα της Ρουμανίας κατά τη διάρκεια της θητείας αυτής. Και για μένα είναι τιμή να εργαστώ σε θέματα που, ε, στα οποία θα εργαστεί η δική μου χώρα, έχοντας την Προεδρία. Ξέρω ότι η κοινή γεωργική πολιτική αποτελεί προτεραιότητα για την Ευρώπη και γι' αυτό σας ρωτώ, κυρία Πρωθυπουργέ, ποιο είναι το όραμα της Προεδρίας της Ρουμανίας και τι προτείνει η Προεδρία σε σχέση με αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα. Σας ευχαριστώ. Κύριος Πρέντα. Ευχαριστώ. Πολύ σύντομα, κυρία Πρωθυπουργέ, του τελευταίου μήνες και εσεί και μέλη τη κυβέρνησή σας άσκησαν κριτική στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και υποστηρίξατε επανειλημμένα ότι η δραστηριότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βασίζεται σε παραπληροφόρηση και σε επιπολαιότητα. Επίσης, και ε, απευθύνεται κριτική στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και είπατε ότι ξένες δυνάμεις ε, ε, το χειραγώγησαν και πώς πιστεύετε ότι μπορείτε να συνεργαστείτε με την Κομισιόν και με το Κοινοβούλιο θεσμικούς εταίρους αφού είπατε ότι δεν πρέπει να υπάρχει εμπιστοσύνη στην Κομισιόν και στο Κοινοβούλιο και το είπατε και στους Ρουμάνους. Και θέλω να σας πω και κάτι ακόμα. Τη στιγμή που συζητάτε για τις προτεραιότητες της Ρουμανικής Προεδρίας, στη Ρουμανία ένα τηλεοπτικό κανάλι διέκοψε την εκπομπή του γιατί ε, τόλμησε να δείξει εικόνες από τη διαδήλωση της 10ης Αυγούστου και είπατε, ε, όπως είπε και ο κύριος Μπουλμέν, ε, δεν υπάρχει ελευθεροτυπία στη Ρουμανία. Θα πρέπει να ανησυχεί αυτό, κυρία Πρωθυπουργέ αν δεν ήσασταν σε μία λογική του Τσαουσέσκου και αν δεν θέλετε να επιστρέψετε στο χρόνο, οπότε η προπαγάνδα ήταν προτιμότερη της αλήθειας ε, και κόβετε το μικρόφωνο του μιλητή. Παρακαλώ, κύριος Ρόνεν, για ένα λεπτό. Μικρόφωνο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι η πρώτη φορά που η Ρουμανία αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου και υπάρχουν πολλά σημαντικά θέματα στα οποία θέλουμε να επιτύχουμε πρόοδο του επόμενου μήνε. Θέλω να τονίσω το θέμα τη οδηγία για την προστασία των καταγγελόντων και είτε αυτοί προέρχονται από τον ιδιωτικό είτε από τον δημόσιο τομέα, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι θα υπάρχουν κανόνε προστασία του. Θα πρέπει να μπορούν να καταγγείλουν τα δικαιώματα ή εγκλήματα που γνωρίζουν. Εάν δεν έχουν εμπιστοσύνη στην ε, προστασία που θα του προσφερθεί, δεν θα περάσουν σε καταγγελίε. Το Συμβούλιο έχει αμφισβητήσει τη νομική βάση της οδηγίας. Όμως, ε, οι νομικές υπηρεσίες του Κοινοβουλίου και του, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν συμφωνούν. Δεν πρέπει λοιπόν να παραμένουμε σε ένα τέλμα στο Συμβούλιο. Ελπίζω ότι η Ρουμανία κατά τη διάρκεια του εξαμήνου της θα κάνει ό,τι μπορεί για να προωθήσει με θετικό τρόπο τις σχετικές διαπραγματεύσεις. Ώστε οι καταγγέλλοντες να έχουν ευρωπαϊκή προστασία με ελάχιστα πρότυπα. Ευχαριστούμε και τώρα... Πού πήγαμε. Κυρία Ταπαρντέλ. Ευχαριστώ, αγαπητοί συνάδελφοι. Η ανάληψη τη Προεδρία από τη χώρα μου αποτελεί πολύ σημαντική στιγμή για τη Ρουμανία και θα αποδείξει η Ρουμανία την διοικητική της ικανότητα και την αξία της, καθώς και το σημαντικό ρόλο που θα παίξει στην διαχείριση των ευρωπαϊκών υποθέσεων και στην ε, οικοδόμηση του μέλλοντος. Θα έχει στρατηγική θέση και θα αποτελέσει ένα δεσμό που ε, θα εναρμονίσει τα διάφορα συμφέροντα που έχουν διαιρέσει την Ανατολική και τη Δυτική Ευρώπη. Νομίζω ότι είναι σημαντικότερο παρά ποτέ σε αυτή την περίοδο της γεμάτη προκλήσεις να δείξουμε ενότητα και αλληλεγγύη για το καλό των Ρουμάνων. Λυπάμαι που σας λέω κύριε Φερχόφστατ, κυρία Κέλλερ και σε άλλου που πήραν το λόγο σήμερα ότι πλανά στα είναι λανθασμένες οι πληροφορίες σας ε, και σας έχουν παραπλανήσει ε, και είναι λυπηρές οι επιθέσεις που κάνετε σήμερα στη Ρουμανία και στην κυβέρνησή της ε, γράφονται στη λογική προεκλογικής εκστρατείας. Η Ρουμανία είναι κράτος δικαίου και η κυβέρνηση της Ρουμανίας υποστηρίζει τις θεμελιώδεις ελευθερίες και τα δικαιώματα των Ρουμάνων ενώ η Προεδρία της Ρουμανίας της, Συγγνώμη, ενώ ε, η δική σα Προεδρία γνωρίζει τι τις αποφάσεις του Συνταγματικού Δικαστηρίου. Ελπίζω ότι το έτος 2019 να είναι ένα έτος χωρίς ελεκτικό μηχανισμό για τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία και να ενταχθούν πλήρω οι δύο χώρε αυτέ στο χώρο Σέγγιν. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και τώρα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο Αντιπρόεδρος της κύριος Άνσιπ. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, κυρία Πρωθυπουργέ, κυρίες και κύριοι βουλευτές, θα να σας ευχαριστήσω όλους για την πολύ έντονη αυτή συζήτηση. Όπως γνωρίζουμε, κατά τη διάρκεια της Ρουμανικής Προεδρίας ε, θα έχουμε το Brexit. Θα έχουμε ευρωεκλογές και τις ε, διαπραγματεύσεις για το επόμενο πι δέλτα πι. Και ταυτόχρονα πρέπει να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις για 242 διαφορετικές προτάσεις. Λοιπόν, θα τα κάνουμε όλα αυτά από κοινού. Μας είπε ο κύριος ε, Γιωχάνης την προηγούμενη εβδομάδα στο Βουκουρέστι, ο πρόεδρος της ε, Ρουμανίας. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής μου εκεί ε, αντιλήφθηκα πως οι Ρουμάνοι υπουργοί τα παίρνουν πολύ στα σοβαρά αυτά. Αναμένω λοιπόν την επικοδομητική συνεργασία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Κομισιόν και της Ρουμανικής Κυβέρνησης κατά τη διάρκεια της Προεδρίας σας και σας εύχομαι κάθε επιτυχία. Σας ευχαριστώ. Μουλτσουμέσκ. Τον λόγο τώρα έχει η κυρία Πρωθυπουργός. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή τις παρεμβάσεις των ε, πρώην συναδέλφων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Για να είμαι ειλικρινής, περίμενα να ακούσω κάποιες προτάσεις, κάποιες λύσεις, μια θετική προσέγγιση, έτσι ώστε οι Ευρωπαίοι πολίτες ε, που σήμερα στρέφονται προς τα μας να δουν απαντήσεις στα προβλήματα που τους απασχολούν απαντήσεις ε, στα εφιστάμενα προβλήματα για διάφορες κοινωνικές κατηγορίες, για διάφορες περιφέρειες και για διάφορες χώρες. Όπως ε, είπα, όταν πήρα το λόγο προηγουμένως, ε, δεν ήρθα να λογοδοτήσω για κάποια πράγματα. Ήρθα εδώ, στο Κοινοβούλιο, ως Πρωθυπουργός μιας χώρας, ως Πρωθυπουργός της Ρουμανίας, για να βρούμε μαζί λύσεις που θα καταστήσουν ισχυρή την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια Ευρωπαϊκή Ένωση που να βρίσκεται πολύ πιο κοντά στους πολίτες όλων των κρατών μελών. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Αντιπρόεδρο για τα καλά του λόγια, για την εμπιστοσύνη που δείχνει η Κομισιόν στην Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Ρουμανίας. Χρειαζόμαστε την υποστήριξή σας και είμαι πεπισμένη ότι από κοινού με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα διασφαλίσουμε την ασφάλεια και τη συνένωση για τους φακέλους και τις προκλήσεις που έχουμε στο Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε κάποια από τα προβλήματα που τέθηκαν. Κυρία Στολοζάν. Οι υπουργοί μας έχουν εμπειρία. Έχουν ασκήσει τη σκιώδη προεδρία και έχουν έρθει σε επαφή τόσο με τις προεδρίες των Επιτροπών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά και με τους ε, επιτρόπους σε σχέση με τα διάφορα ζητήματα και φακέλους. Σίγουρα υποστηρίζουμε την, ε, μας υποστηρίζει και η Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου ήθελα να μην θεωρήσετε ότι οι υπουργοί δεν θα χειριστούν τους φακέλους ή δεν θα μπορέσουν να δώσουν θετικές απαντήσεις στα προβλήματα που έχουν επιλύσουν. Από τη δική σας πλευρά αναμένω να έχετε εμπιστοσύνη στους υπουργούς της Ρουμανίας και στην ικανότητα της Ρουμανίας. Αναφερθήκατε στην υποχρέωση της ε, Πρωθυπουργού να συναντηθεί με τους Πρωθυπουργού της Γαλλίας ή των κατοχωρών. Είμαι ανοιχτή στο να το κάνω αυτό, είμαι ανοιχτή στο να μεταβώ στο Ολλανδικό Κοινοβούλιο και στο να διαβιβάσω στον πρόεδρο, τον πρόεδρο της ε, Ρουμανίας να προσεγγίσει αυτά τα θέματα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, γιατί ο πρόεδρος συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Σε ό,τι αφορά τώρα την Ευρωζώνη, το Δεκέμβριο του 2018 ε, ορίσαμε το έτος ε, ότι θα μπούμε στο ευρώ και πρέπει να κάνουμε κάποια βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Όμως, εμείς έχουμε κρατήσει το λόγο μας και αν θέλετε το πρόγραμμα αυτό είμαστε στη διάθεσή σας να σας το παρουσιάσουμε. Ευχαριστώ τον ε, πρόεδρο της Ομάδας Σοσιαλιστών και Δημοκρατών ε, για την υποστήριξη και του εγγυόμαστε ότι υποστηρίζουμε το κράτος δικαίου. Ταυτόχρονα σεβόμαστε και τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά και τα δικαιώματα όσων έχουν υποφέρει λόγω λανθασμένων αποφάσεων της δικαιοσύνης. Κύριε Φερχόφστατ, λυπάμαι ε, που έφυγε ο κύριος Φερχόφστατ από εδώ. Θέλω να τον διαβεβαιώσω ότι εμείς γνωρίζουμε τους φακέλους και τις προκλήσεις ε, που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Ακριβώς γι' αυτό ζήτησα συνένεση, γιατί χρειαζόμαστε τη συναπόφαση, χρειαζόμαστε τη συνένεση και θα εργαστούμε προς την κατεύθυνση αυτή. Ταυτόχρονα, περίμενα ότι ένας επικεφαλής ε, πολιτικής ομάδας ε, να κάνει κάποιες παρατηρήσεις σε σχέση με το ευρωπαϊκό θεματολόγιο. Όχι να κάνει παρατηρήσεις για τα ιστορικά προβλήματα μιας χώρας που μόλις ανέλαβε την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για λόγους αξιοπιστίας νομίζω ότι θα πρέπει να μιλάει κανείς γνωρίζοντας ε, τα γεγονότα. Και θα ήθελα να μου πει ο κύριος Ερχόστατ σε τι έχει να επιπλήξει τη ρουμανική κυβέρνηση τι καταλογίζει και ταυτόχρονα ζητώ από τον κύριο Φερχόφστατ να αφήσει τους Ρουμάνους να αποφασίσουν μόνοι τους ε, να μην προσπαθεί να παρουσιάσει τις δικές του πεπιθήσεις ε, στους Ρουμάνους, να μην προσπαθεί να περάσει τις δικές του πεπιθήσεις στους Ρουμάνους. Είμαι πεπισμένη ότι οι συνάδελφοί μου θα παρουσιάσουν προτάσεις ε, για τις άλλες χώρες, όμως θα πρέπει να αφήσουμε τον κάθε λαό και τους πολίτες της κάθε χώρας ε, να ε, επιλέξουν ε, και να δράσουν βάσει των δικών τους πεπιθήσεων. Κύριε Κέλλερ. Είπατε ότι χιλιάδες Ρουμάνοι βγήκαν στο δρόμο για να ζητήσουν μια καλύτερη διακυβέρνηση. Νομίζω ότι δεν ενημερωθήκατε σωστά. Θα ήθελα να σας δώσω κάποια αριθμητικά στοιχεία που δείχνουν ε, τι σημαίνει καλή διακυβέρνηση στη Ρουμανία. Έχουμε οικονομική ανάπτυξη πάνω από 4%. Το έλλειμμά μας ε, είναι 2,96%. Ενεργεία κάτω από 4%. Οι επενδύσεις στη Ρουμανία αυξήθηκαν πάνω από 10%. Και πιστεύω αυτό σημαίνει καλή διακυβέρνηση. Και πιστεύω ότι η παραπληροφόρηση κάποιων συναδέλφων ε, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, οδήγησε σε αυτή την αντίληψη. Αν θέλετε μπορώ να σας στείλω όλα τα αριθμητικά στοιχεία και όλα όσα έχει κάνει η κυβέρνηση της Ρουμανίας για να διαβεβαιώσει την βελτίωση του επίπεδου διαβίωσης και μια καλή διακυβέρνηση για τη Ρουμανία και τους Ρουμάνους. Πιστεύω ότι θα πρέπει να συγκρίνετε και με τα αποτελέσματα άλλων χωρών και τότε θα καταλάβετε ότι η Ρουμανία έχει μια κυβέρνηση η οποία ξέρει τι πρέπει να κάνει και η οποία έχει ασχοληθεί με τα προβλήματα των Ρουμάνων και της Ρουμανίας. Ο κύριος Πάξας ε, μας ε, ρώτησε γιατί ε, το ενδιαφέρον για την Ένωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντικαταστάθηκε με τη διαίρεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω ότι είναι μια ερώτηση που πρέπει να τη θέσουμε όλοι μα Νομίζω ότι πρέπει να εργαστούμε περισσότερο και να δούμε τι μας ενώνει και να δούμε και να εκτιμήσουμε λιγότερο αυτά που μας χωρίζουν. Γιατί μόνο αν είμαστε μαζί ενωμένοι, μόνο μέσω της συνοχής, μπορούμε να κάνουμε σημαντικά βήματα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Μαρία Ζωάο για τα πολύ καλά της λόγια. Πράγματι, η Σύνοδος Κορφής στο Συμπίου θα μας δώσει την ευκαιρία μαζί να χαράξουμε το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιστεύω ότι μίλησε για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το να μιλάμε, συγγνώμη, για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης σημαίνει να βρίσκουμε μαζί, ανεξάρτητα της πολιτικής μας ομάδας, ε, την καλύτερη δυνατή λύση που να είναι κοντά στους πολίτες, έτσι ώστε να έχουμε ένα κοινό και το καλύτερο δυνατό μέλλον για τους πολίτες της Ένωσης. Κύριε Χόκμαρ, και η κυβέρνηση θα πρέπει να καταπολεμήσει τη διαφθορά. Πολλές φορές ε, το έχω πει. Δεν έχουμε κανένα νομοθέτημα επιτάπητο στο τραπέζι της κυβέρνησης που αναφέρεται στην αμνηστία. Δεν θέλουμε να υπερασπίσουμε κανένα, θέλουμε μόνο να προστατεύσουμε τους πολίτες των οποίων έχουν καταπατηθεί τα δικαιώματα. Και θα χαιρόμουν πάρα πολύ όταν, μιλάμε για το κράτος δικαίου, όταν μιλάμε για δικαιοσύνη, όλοι να αγωνιστούμε κατά της διαφθοράς. Και η κυβέρνηση της Ρουμανίας θα το πράξει αυτό. Όμως ε, ταυτόχρονα να προστατεύσουμε και τα δικαιώματα των πολιτών που έχουν πληγή από αποφάσεις της δικαιοσύνης, από τα μυστικά πρωτόκολλα συνεργασίας μεταξύ της δικαιοσύνης και των μυστικών υπηρεσιών. Αυτοί που τώρα φωνάζουν δυνατά και δηλώνουν ότι αγωνίζονται κατά της διαφθοράς, ότι θέλουν να αγωνιστούν υπέρ του κράτους δικαίου, πολλοί από αυτούς θα κρύψουν τι συνέβη στην πραγματικότητα στη Ρουμανία. Και μάλιστα ήταν μέρος αυτού του συστήματος που οδήγησε στην ε, καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Κύριε Μαρινέσκου, η δική σας θέση κατά της κυβέρνησης της Ρουμανίας είναι αδικαιολόγητη. Είπατε ότι υπήρξαν επιθέσεις στην κυβέρνηση, ε, της κυβέρνησης συγγνώμη, κατά της δικαιοσύνης. Εγώ δεν θυμάμαι και κανείς ούτε ένας Ρουμάνος πολίτης ε, δεν νομίζω ότι μπορεί να πει ότι η κυβέρνηση της Ρουμανίας έλαβε κάποια απόφαση κατά της δικαιοσύνης. Όλοι οι νόμοι που αναφέρονται στη δικαιοσύνη ψηφίστηκαν στο Κοινοβούλιο της Ρουμανίας και το Ρουμανικό Κοινοβούλιο εκφράζει την ψήφο των Ρουμάνων πολιτών. Μιλήσατε για ευρωπαϊκά κονδύλια, για ευρωπαϊκά ταμεία. Νομίζω ότι αναφερόσασταν στην τεχνοκρατική κυβέρνηση, γιατί εμείς κατά την ε, δική μας περίοδο διακυβέρνησης ε, μέσα σε ένα χρόνο ε, ανακτήσαμε τα ποσά, έχουμε πολύ καλή απορρόφηση των κονδυλίων ε, για να μην μιλήσουμε για το τι συμβαίνει στον τομέα της γεωργίας, είναι το 27% που είναι ο ευρωπαϊκός μέσος όρος. Εγώ πιστεύω ότι ε, το γεγονός ότι η κυβέρνηση αυτή υποστηρίζει τους πολίτες έχει αποδεικτεί από τα μέτρα που υιοθετούμε και όχι από αυτούς που ψήφισαν εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά της ίδιας τους της χώρας. Κυρία Μπρέσο, πράγματι η εδαφική σύγκληση είναι πολύ σημαντική και δεν πρέπει να αφήσουμε να καθυστερήσει καμία περιφέρεια. Εμείς ε, όλες τις προτάσεις σας θα τις δεκτούμε με ανοιχτό πνεύμα για να προωθήσουμε το θέμα αυτό στο θεματολογιό μας. Είπατε ότι 20 εκατομμύρια νέοι θα ψηφίσουν για πρώτη φορά και τι μπορούμε να κάνουμε για να τους πείσουμε να έλθουν στις κάλπες. Καταρχήν, θα πρέπει να δείξουμε ότι έχουμε λύσεις για αυτούς. Δεύτερον, θα πρέπει να δείξουμε ότι η δική μας διένεξη δεν είναι μεταξύ πολιτικών ομάδων, μεταξύ πολιτών του ίδιου κράτους μέλους, αλλά ότι οι δικές μας διαφωνίες και οι δικές μας λύσεις είναι για αυτούς. Ότι μπορούμε να φέρουμε προσθέμενη αξία και ότι αυτοί θα πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο των αποφάσεων που λαμβάνουμε στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Και έχω την πεποίθηση ότι μαζί μπορούμε να το πράξουμε αυτό. Έχω εμπιστοσύνη στους Ευρωβουλευτές, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο Συμβούλιο, ότι μαζί θα μπορέσουμε το επόμενο εξάμεινο να δώσουμε τις απαντήσεις που περιμένουν αυτά τα 20 εκατομμύρια νέων, τις απαντήσεις που περιμένουν τα 500 εκατομμύρια πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κυρία Γιάροκα, ελπίζω να μην θα σημαίνω το όνομά σας. Μας είπατε ότι είμαστε ένα φτωχό κράτος και θα, πρέπει να κάνουμε κάτι προς αυτή την κατεύθυνση. Το τελευταίο έτος ακριβώς αυτό κάναμε. Έχουμε βελτιώσει το επίπεδο διαβίωσης. Είδαμε ότι η λιτότητα δεν αποτελεί λύση για τη χώρα μας, ούτε και για άλλα κράτη-μέλη. Ε, αυξήσαμε τους μισθούς, αυξήσαμε τις συντάξεις, αυξήσαμε τους μισθούς των γιατρών ε, και των ε, εκπαιδευτικών αυξήσαμε τα επιδόματα για τους ευπαθείς πληθυσμούς και ε, προσθέσαμε το περιβάλλον και νομίζω ότι όλα αυτά θα πρέπει να τα κάνουμε για να μην μιλάμε για ανέχεια πέρα από τις αποφάσεις που πρέπει να λάβουμε από κοινού σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και σε σχέση με την τελευταία ερώτηση, θέλω να απαντήσω στις τελευταίες κατηγορίες. Σκέφτηκα πολύ αν αξίζει ή δεν αξίζει να δώσω την απάντηση αυτή. Όμως εγώ πιστεύω ότι ως πολίτες θα πρέπει να κάνουμε μια διαφοροποίηση μεταξύ μιας εχθρικής συμπεριφοράς και μια ανοιχτή συμπεριφοράς. Κύριε Πρέντα, η κυβέρνηση της Ρουμανίας και ο Πρωθυπουργός, ή Πρωθυπουργός της Ρουμανίας δεν επικρίνουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εγώ ήμουν